και από την Επιτροπή ΕΚΟΝ για να μην υπάρξουν αντιρρήσει για μια πράξη εξουσιοδότηση η οποία ανακοινώθηκε στην έναρξη τη χθεσινή συνεδρίαση. δεν κατατέθηκαν λοιπόν τέτοιε καταγγελίε και ενστάσει εντό τη χρονική προθεσμία 24 ώρων που εξαπνεύσε στις 5 και 15. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παραγραφός 6 του κανονισμού, η σύσταση λοιπόν θεωρείται εγκεκριμένη και θα δημοσιευθεί με τα ε, εγκεκριμένα κείμενα αύριο, Τετάρτη 5 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.